Okay. Dear colleagues, ladies and gentlemen, let... Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ας ξεκινήσουμε. Και πριν ε, ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη, πρέπει να κάνω μια ανακοίνωση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Νομίζω έχει σημασία για τις πολιτικές ομάδες. Τα 23, 24 και 25 Μαρόκο αναβάλλονται. Το Μαρόκο λοιπόν δεν θα το συζητήσουμε σήμερα. Για το σημείο 26 λοιπόν Κεντρική Αμερική Συμφωνία Σύνδεσης θα πρέπει να έχουμε παρόντες τους πάντες την ώρα που θα ολοκληρώνεται το 22 δηλαδή στις 10.40 λίγο πολύ για να μην ε, χρειαστεί να περιμένουμε μία ώρα. Ελπίζω να είναι σαφές το μήνυμα. Διάλειμμα δεν θα γίνει μετά το σημείο 22. Θα περάσω απευθείας στο σημείο 26 και ας φροντίσουν οι πάντες να ενημερωθούν και βέβαια και ο εισηγητής του 26. τούτου λεχθέντος. Ξεκινώ με την ημερήσια διάταξη και το σημείο 15. Προσχώρηση της ΟΜΟΑ στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρική σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφενός και των κρατών του Ειρηνικού αφετέρου με τον David Μάρτιν εισηγητή. Πριν όμως του δώσω το λόγο θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, κύριο πρεσβευτή της ε, ε, ΣΑΜΟΑ, κύριο Φατουμανάβα. Πάλου Τερό και ζητώ συγγνώμη για την προφορά. Δεν νομίζω ότι είχε καμία σχέση με την προφορά του ονόματός σας αυτό που είπα, αλλά καλώς ήρθατε όπως και να έχει. David Μάρτιν, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και καλώς ορίσατε κύριε Ξέρετε ότι είχα αναλάβει την έκθεση για το προενταξιακό μέσο τη, με τον ειρηνικό στην προηγούμενη θητεία το 2011 έπρεπε να εγκριθεί, το είχα υποστηρίξει αναφανδόν. Ε, περιμέναμε ένα πλήρες προενταξιακό μέσο να προκύψει από αυτή τη συμφωνία Δυστυχώς όμως μετά την αποχώρηση της Παπουάς Νέαχους Γουινέας το 2015 από τη συμφωνία διακόπησαν οι συνομιλίες για το πρωταξιακό μέσο ΙΠΑ και αν δεν μας ε, επιφυλάσσει καμία έκπληξη η Επιτροπή σήμερα το πρωί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι καινούριο για το μέλλον. Μακάρι να συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα ήταν το ιδεώδες. Ε, αποτελεί λοιπόν ένα μέσο ανοιχτό για προσχώρηση ε, και σε άλλα κράτη και η Σαμόα θέλει να, αξιολογεί, να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία. Είναι στο σύστημα τα πάντα πριν όπλων, στο προτιμησιακό σύστημα, που όμως θα λήξει, μετά τη μετα... θα εκπνεύσει μετά την ε, ε, εκπνοή της μεταβατικής περίοδου και θα αρχίσει να ισχύει για τη Σαμόα το πιο γενναιόδωρο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, ενώ θέλει να διατηρήσει την ε, αδασμολόγητη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές. Από 1η Ιανουαρίου του 2019, εάν δεν, γίνει αυτή, αν δεν δοθεί αυτή η παράταση, θα διαταραχθεί η εταιρική σχέση της ΣΑΜΟ. Έχουμε να κάνουμε με εξαγωγές της τάξης των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ σε τιμές του 2017, μικρό για τα, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά πάρα πολύ σημαντικό ποσό και όγκο συναλλαγών για ένα κράτος μικρό όπω η Σαμόα. Και επιπλέον των προτιμήσεων ε, θα έχουμε με την ενδιάμεση αυτή συμφωνία την ε, δυνατότητα να εγκαθιδρυθούν μακρο πρόθεσμα σχέσει εταιρικέ ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση που πιστεύουμε ότι θα οδηγήσουν και σε μεταρρυθμίσεις και σε πιο μακροχρόνιες επενδύσεις. Έτσι, ανταλλαγή ε, ε, εμπορευμάτων σε συμμετρικούς όρους με αδασμολόγητη πρόσβαση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και 8,2 εκατομμύρια όγκο συναλλαγών υπό απελευθέρωση από τη ΣΑΜΟΑ για περίοδο 20 ετών θα είναι μία η μία εκδοχή, η μία πτυχή αυτής της συμφωνίας, ε, αγαθά τα οποία αποκλείονται είναι τα προϊόντα αλληλείας, ε, ε, εμφαλιωμένο είδωρ λοιπά, μεταλλικό είδωρ κτλ. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις για την Σαμόα, χωρίς να είναι όμως ιδιαίτερα φιλόδοξες αυτές οι προβλέψεις, ε, μια στήριξη για την βιώσιμη ανάπτυξη επιπλέον θα χρειαστεί. Έχουμε μια ρήτρα μη εκτέλεσης για τη Συμφωνία Κοτονού ε, που κατά κάποιον τρόπο θα αποτελούσε ένα μηχανισμό ελέγχου της εφαρμογής που όμως εκπνέει και αυτή το 2020. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να ε, επανεξεταστούν αυτές οι λοιπές συμφωνίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν να ενταχθούν στο τέλος κάποια στιγμή σε, μια ολοκληρωμένη, σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο. Ε, μέσα από το πρόεδρο μέσο. Θα σταματήσω εδώ γιατί έχω και άλλα πράγματα να πω, αλλά ας μιλήσει ο κύριος Προσευτής πρώτα. Ο Πρόεδρος ευχαριστώ πολύ και οδησηγητέ ο κύριος Γουάς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Είμαι σκιώδη ηγητή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο στην υπόθεση αυτή και θα ήθελα να κάνω κάποιε παρατηρήσει. Καταρχά, είμαστε ενώπιον μια ε, πρόταση ε, για προσχώρηση τη ΑΜΟΣ αυτήν την εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, ειρηνικού, κάτι που ξεκίνησε με την ε, Παπουανέα Γουινέα, της νήσους Φίτζη και μπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση ενός ε, εμπορικού πλαισίου συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των συναλλαγών. 0,1% του παγκοσμίου όγκου εμπορικών συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αντιστοιχούν σε αυτές τις συναλλαγές. Η Σαμόα δεν υπάγεται πλέον από το 2014 και μετά στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και άρα δεν μπορεί να ωφελείται πλέον από το σύστημα γεννητικευμένων ε, προτιμήσεων. Από φέτος το Δεκέμβριο δηλαδή λύγει το σύστημα αυτό για την ε, Σαμόα. Για να μπορέσει να έχει τα ωφέλη της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά θα ήταν πολύ σημαντικό να δεχθεί την, το αίτημα αυτό για προσχώρηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού αυτή η προσωρινή εταιρική σχέση ήδη έχει προβλεφθεί για δύο άλλα κράτη. Έχουμε να κάνουμε με συμφωνίες τελευταία ανάλυση, οι οποίες ε, στοχεύουν στην υποστήριξη της ανάπτυξης ε, των ε, χωρών που αφορούν και πέραν ε, διαφόρων κανόνων για το εμπόριο και φυτογίνων ε, μέτρων πρέπει να εξασφαλίζουν και μέτρα με δυνατότητα πρόσβασης ε, στις αγορές ασύμετρες για συγκεκριμένα προϊόντα και με διευκόλυνση δυνάμει του άρθρου 108 και του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε να κάνουμε εδώ λοιπόν με μια συμφωνία εμπορική που θα προτιμούσαμε να ήταν πολύ πληρέστερη και να συνοδεύεται ή να εντάσσεται μέσα σε μια στρατηγική που θα φορούσε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχέσεών της με τις χώρες ΑΚΕ μετά το 2020. Συμφωνώ λοιπόν ότι θα πρέπει οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης ε, να ε, συνδεθούν με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία των Παρισίων τι μεγάλες αυτές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο εμείς όσο και οι χώρε του ειρηνικού. Thanks a lot. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Τζουρτ Κερτοντάλ. Ευχαριστώ πολύ. Μια σύντομη ερώτηση. Έχω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κύριο Πρέσβη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Έχουν προχωρήσει οι εξελίξεις ε, από τότε που ε, συμφωνήσαμε για την διάμεση συμφωνία για το προεταξιακό μέσο, όπως είπε και ο Ντέιβιτ. Στην περασμένη θητεία έχουμε αλλάξει τώρα συμφωνίες για την βιώσιμη ανάπτυξη και την ε, οικονομική εταιρική σχέση. Είναι πολλές επικρίσεις που ακούγονται στο Κοινοβούλιο για το ε, γεγονός ότι είναι μικρές αναφορές στη βιώσιμη ανάπτυξη και απλώς υπάρχει μια σύνδεση με τη Συμφωνία ε, Κοτονού. Μετά όμως ε, από τις συζητήσεις που είχαμε στο Κοινοβούλιο είδαμε ότι έχουν προγραμματιστεί κάποιες συζητήσεις που έχουν γίνει με την Κάνα, με την αρχή Ελεφαντοστού Υπάρχουν κάποια σχέδια ε, στις χώρες της Αφρικής για συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, παρόλο που δεν τα αναφέρουν ρητά οι συνθήκες και οι συμφωνίες. Και στο προσωρινό προενταξιακό μέσο, το ξέρω ότι την αναφέρεται, αλλά έχετε βάλει καμία προσπάθεια να συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών στην ε, όλη αυτή η προσπάθεια και τον προβληματισμό για την βιώσιμη και η φόρο ανάπτυξη και εμπόριο. Uh, το είπα, προφανώ είναι η Συμφωνία Οικονομική Σχέσης. Σχέση και όχι το πρώτο εξέχω. Ε, είμαι σκιώδη τη της ε, ΔΕΒΕ, της ε, Επιτροπής Ανάπτυξης, για την συμφωνία αυτή την εμπορική με τη ΣΑΜΟΑ τη Δευτέρα. είχαμε μια πρώτη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Τα έχω πει και στον πρέσβη τον οποίο και καλωσορίζω εδώ, έχω κάποια επιφυλακτική θεώρηση εγώ. Το πρώτο έχει να κάνει με τη Συμφωνία των Παρισίων. Όλοι είδαμε την ε, έκθεση των εμπειρογνώμων για το κλίμα που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, οι οποίοι μας είπαν ότι όχι απλώς πηγαίνουν ε, άσχημα τα πράγματα, αλλά θα πρέπει να επιταχύνουμε τη δράση μας. Και οι κύριοι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιοι άλλοι και τα μεγαλύτερα θύματα είναι τα νησιωτικά κράτη όπως είναι η Σαμόα και κάποια άλλα. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε το θέμα του εμπορίου γιατί το διεθνές εμπόριο ευθύνεται για το 1 πέμπτον των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα παγκοσμίω. Οπότε οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο ε, για εφαρμογή των συνθήκων του ε, Παρισιού εργαλείο είναι το εμπόριο, δεν είναι αυτός ο σκοπός για να φτάσουμε στους στόχους αυτούς, οι οποίοι είναι σημαντικότεροι. Γι' αυτό είναι αρκετά απορία άξιο, όπως είπαν και οι συνάδελφοι προηγουμένως, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διατάξεις για την εφόρο ανάπτυξη, σχετικό κεφάλαιο, που κανονικά όλα αυτά είναι δεσμευτικά, υποχρεωτικά και εκτελεστέ. Το κοτονού σημαίνει διάλογο. Πολύ ωραίο είναι ο διάλογος, αλλά αυτά δεν είναι υποχρεωτικά και ε, δεσμευτικά που θα πρέπει να επιβάλλονται, ας πούμε, και ε, από τον νόμο για ένας ε, μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Επίσης δεν, προσ... δεν προβλέπεται και δημιουργείται και κακό προηγούμενο. Την περασμένη εβδομάδα εμείς ψηφίσαμε ότι είμαστε υπέρ συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις επιχειρήσεις ε, συνθήκη δεσμευτική. Όπως έχουμε δει στο κλάδο της ένδυσης ε, που υπάρχουν ε, δεσμευτικές και υποχρεωτικές διατάξεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο διεθνές εμπόριο. Είναι και έκθεση συναδέλφου Χάουταλα. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε και εδώ συνέπεια και να προσαρμόσουμε και τη συγκεκριμένη εμπορική συμφωνία στους κανόνες. Αναβολή δεν χωράει. Μα το είπαν και οι εμπεργνώμονες για το κλίμα. Δεν έχουμε χρόνο. Τώρα πρέπει να γίνει αυτό. Και δεν μπορούμε να δεχτούμε ε, συμφωνία χωρί κεφάλαιο για η φόρο ανάπτυξη. Πράγματι δεσμευτικό. Κάτι άλλο που δεν ακούσαμε. Είναι σε ένα μαύρο κατάλογο, μαύρη λίστα η Σαμόα μη συνεργαζόμενη χώρα σε θέματα φορολογικά. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να αναθεωρηθεί αυτό. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε επαφή με τη Σαμόα, αλλά γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα θέματα αυτά. Έχουμε δύο ψηφίσματα τουλάχιστον σχετικά και το ένα λέει ότι θα ζητηθεί αναστολή της συμφωνίας αν δεν συνεργάζεται η χώρα και αν δεν βγει από το μαύρο κατάλογο δεν μπορούμε να ε, συνεχίζουμε τη συνεργασία μας σε άλλα θέματα. Το έχω συζητήσει με τον πρέσβη. Είπε ότι η χώρα κάνει ό,τι μπορεί για να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και αυτό θα πρέπει να ενταχθεί στη συμφωνία και όχι να αναβληθεί εκ νέου. Αυτά είναι δύο σημαντικά σημεία και θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε και να λήξουν πριν υπογραφεί η συμφωνία γιατί το ζητάει ο κόσμος, οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εμπορικές συμφωνίες να πηγαίνουν προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά και είναι και προς το καλό της ΣΑΜΟΑΣ. γιατί αυτοί που θα πληθούν, πληγούν περισσότερο από την αύξηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα είναι οι συνάδελφοι και οι φίλοι των νησιωτικών κρατών, όπως είναι η Σαμόα. Σας ευχαριστώ. Έχω κι εγώ μια ερώτηση και για τον πρέσβη και για την Επιτροπή. Τον τελευταίο καιρό έχω ακούσει για μια συζήτηση για εξόριξη πετρελαίου στη, στον ωκεανό, στην περιοχή, για γεωτρήσεις. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν αυτό το ζήτημα και της εξαγωγής των προϊόντων που θα, που θα εξορίσονται σε μεγάλα βάθη αν, αν εντάσσεται στην ΕΠΑ, στην Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας και εάν αυτό εφορά κάποια περιοχή που να είναι στα χωρικά ύδατα της Σαμόα και αν ναι, έχει γίνει κάποια αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου Λοιπόν, κύριε Πρέσβη, έχετε το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ετέθησαν και μετά θα μιλήσει η Επιτροπή. Κύριος Πρέσβης. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να κάνουμε μια σύντομη δήλωση σε σχέση με την αίτηση της ΣΑΜΟΑ να ενταχθεί στο υφιστάμενο όργανο συνεργασίας, συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών του Ειρηνικού. Η ΣΑΜΟΑ θεωρεί ότι το διεθνές εμπόριο είναι ουσιαστικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και την καταπολέμηση της, και εξάλληψη της φτώχειας. Ο τελευταίος στόχος είναι πολύ κρίσιμος και στην καρδιά των εταιρικών σχέσεων με τις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες ΑΚΕ. Είμαστε μία από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ανάμεσα στις χώρες ΑΚΕ. Και επίσης γνωρίζουμε ε, και βιώνουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης και τις μενουμερούς προσέγγισης στη διπλωματία, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα της ανθρωπότητας. Κύριε Πρόεδρε, η χώρα μου δεν θα είχε συμφέρον να ενταχθεί σε μια εμπορική ή άλλη συμφωνία η οποία να έθετε σε κίνδυνο την επιβίωση της χώρας. Θεωρούμε ότι αυτή η Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας είναι εργαλείο που θα υποστηρίξει τις προσπάθειες που κάνουμε για βελτίωση της κατάστασης της οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις μας και θα εμβαθύνει τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχέσεις που μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών του Ιωνικού είναι ήδη ισχυρέ. Θα μας δώσει την εδατότητα να έχουμε μια ουσιαστική εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε ανοιχτή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά για τα προϊόντα από την Σαμόα, δεδομένου ότι δεν θα μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας έδινε μετά το 2018 η Συμφωνία ε, τα πάντα πληνόπλων. Οι φυσικές καταστροφές, τσουνάμι και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν καταγραφεί και έχουν φανεί τι καταστροφικές επιπτώσεις μπορούν να έχουν και πόσο αυτά θα επιδεινωθεί ε, πρόσφατα το νότιο, το 2009 μάλιστα, το, το νότιο μέρος της χώρας μου καταστράφηκε από τσουνάμι. Το λέω αυτό γιατί η πρόσβαση στην αγορά δεν αρκεί από μόνη της. Χρειάζεται βεβαίως να μπορεί κανείς να συμμετέχει στο διεθνές εμπόριο με ανταγωνιστικότητα και η Διεθνή Συμφωνία είναι στοιχείο αυτού του στόχου. Η συμφωνία αυτή θα δώσει τη δυνατότητα και σε ευάλωτε ομάδες, ιδιαίτερες ομάδες όπως η νεολαία, όπως οι γυναίκες να συμμετάσχουν ενεργά στην οικονομική ζωή. Η συμμετοχή των νέων και των γυναικών έχει ε, προβλεφθεί στις δομές που δημιουργούμε για τη διαχείριση αυτής της συμφωνίας. Είναι εξάλλου η συμμετοχή αυτών των ανθρώπων στοιχείο του τρόπου ζωής μας. Θα μπορέσει λοιπόν αυτέ αυτές οι επιτροπές, αυτές οι ομάδες παρακολούθησης να συμμετάσχουν και να προκαλέσουν πραγματικές αλλαγές. Είναι πλήρως ενταγμένες και συνδεδεμένες με τα συμβούλια των ε, χωριών, της τοπικές μας κοινωνίας. Οι δυνατότητες, οι ευκαιρίες που θα ανοίξουν ε, για αυτές τις ε, περιφέρειες, αγροτικές περιοχές, έχουν τεράστια σημασία γιατί θα δώσουν τη δυνατότητα για κοινωνική κινητικότητα, για ανέλυξη κοινωνικά, να καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, θα βοηθήσουν τις γυναίκες. Θα, θα συνεισφέρει ουσιαστικά επίσης αυτή τη συμφωνία στην... Ε, στις εθνικές μας στρατηγίες για την ανάπτυξη. Έχουμε κάνει διαβούλευση και θα κάνουμε διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους, όμως τελικά την δύσκολες αποφάσεις οφείλει να τις λαμβάνει η κυβέρνηση και να λογοδοτεί για αυτές, μιας και αποτελεί την εκτελεστική εξουσία στη χώρα. Σε συνεργασία βεβαίως με την νομοθετική εξουσία και τη δικαστική εξουσία. Η ΣΑΜΟΑ θεωρεί ότι η εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΑΚΕ είναι έχει, ε, έχει ένα θέμα, μάλλον από ένα κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη και συγκεκριμένο άρθρο το 15 για τα εργατικό δίκαιο. Η Σαμόα θεωρεί ότι αυτές οι υφιστάμενες προβλέψεις θα κατευθύνουν και θα σχηματοποιήσουν τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο μέλλον. προσπαθήσω τώρα να απαντήσω σε ένα θέμα που ετέθη, το φορολογικό καθεστώς, το οποίο έχει σχετιστεί, μάλιστα έχει συνδεθεί με την δυνατότητα της ΑΜΟΑ να ενταχθεί σε αυτή την οικονομική συνεργασία. Δηλώνω ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να λυθεί το θέμα. Έχω συζητήσει το θέμα πολλές φορές με άλλους πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τότε που η Σαμόα εντάχθηκε σε αυτή τη μαύρη λίστα πέρυσι τον Οκτώβριο. Ε, στις 23 Νοεμβρίου μάλιστα θα οργανώσουμε διάσκεψη για το θέμα προσπαθώντας να καταδείξουμε ότι η Σαμόα επιθυμεί τη συνεργασία με την ομάδα ε, καλών πρακτικών βελτιστής συμπεριφοράς του Συμβουλίου. Αυτός ο κώδικας καλής συμπεριφοράς υιοθετείται από την Σαμόα. Θεωρούμε ότι το θέμα αυτό μπορεί να επιληθεί με τρόπο ικανοποιητικό και για τα δύο μέρη τους επόμενους μήνες. Η Σαμόα θεωρεί ότι οι αρχές με βάση τις οποίες καταρτίζεται αυτός ο κατάλογος, αυτή η μαύρη λίστα, θα πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις, όχι μόνο στις χώρες εκεί, αλλά ακόμα και σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΣΑΜΟΑ προσπαθεί να ενταχθεί σε μια υφιστάμενη εμπορική συμφωνία που έχει ήδη καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχοντας και στο PNG και στο FNG, προσπαθώντας να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών μας, να ενταχθούμε στο παγκόσμιο σύστημα και να βελτιώσουμε ιδιαίτερα τη ζωή των ευάλωτων ομάδων, των νέων και των γυναικών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την προσοχή σας και για τη δυνατότητα που μου δώσατε να παρευρεθώ εδώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Πρέσβη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρία Σκόλα. Thank you, Πρόεδρε, ευχαριστώ. και κύριοι αξιότιμη πρεσβευτά τη ΣΑΜΟΑ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα θέματα που έχουν επισημανθεί εδώ. Είναι όντως μικρό και το νησιωτικό κράτος η ΣΑΜΟΑ. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να την ενσωματώσουμε σε αυτή την εταιρική σχέση. Ο, εισηγητής, ο εισηγητής έχει επισημάνει πολύ σωστά ότι η διαπραγμάτευση έγινε πριν από περισσότερα από 10 χρόνια και εντωμεταξύ έχουν λάβει χώρα αρκετέ ε, αλλαγές στην πολιτική, κυρίως για το εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη. Τα προενταξιακά μέσα πάντω είναι ευέλικτα ε, εργαλεία, μπορούν να Οι εταιρείε οικονομική εταιρική σχέση, συγγνώμη, είναι ευέλικτα μέσα, μπορούν να Ε, μπορούν να προβλέψουν δηλαδή και κυρώσεις και ε, συνέπειες αν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις και τα Τώρα έχουμε την ε, κίνηση των συνομιλιών για το πλαίσιο μετά Κοτονού. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει ιδιαίτερος για σαφείς διατάξεις, σκληρές διατάξεις και στην υπόθεση αυτή του Κοτονού. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα με μια δομή συμφωνιών. Έχουμε δηλαδή τη συμφωνία πλαίσιο που ορίζει τα, ε, το γενικό πλαίσιο και τις ε, επιμέρους ε, και εν επιμέρους πλαίσιο μέτρων μέσα στο οποίο έρχεται να ενταχθεί αυτό το, αυτή η <laughs> Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης. Έχουμε ένα θέμα με τα δικαιώματα των εργαζομένων που προβλέπονται ήδη από την οικονομική εταιρική σχέση. Προβλέπεται ήδη ότι θα αναπτυχθεί ένα φόρουμ διαλόγου. Ε, η ΣΑΜΟΑ ως παρατηρητής ήδη συμμετέχει με την Παππούα Νέα Γουινέα και τα Φίτζη, τους ε, τωρινούς μας εταίρους. 24 Οκτωβρίου προβλέπεται προσεχής ε, σύνοδος εδώ στις Βρυξέλλες με θέμα θέματα όπως την, ε, το θεματολόγιο για τη βιωσμία ανάπτυξη, την αλία, το περιβάλλον, τα εργασιακά δικαιώματα, και ένα θέμα το οποίο θα έχει να κάνει με τις μη συνεργαζόμενες φορολογικές δικαιοδοσίες. Επομένως μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον φόρουμ διαλόγου αυτό το μέσο της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης. Μπορεί να μας βοηθήσει να ενισχύσουμε την επιρροή μας, αλλά και να προβάλλουμε τις αξίες μας σε περιοχές που ξέρουμε ότι κατά τα άλλα είναι υπό την αιγίδα λίγο πολύ άλλων μεγάλων παραγόντων όπως η Κίνα, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία. Θέλουμε κατά τα άλλα, εμείς από πλευράς μας, να έχουμε ο, εγκάρσιες διατάξεις, ομοιόμορφες διατάξεις σε όλα τα μέσα αυτά και για όλους τους τομείς. Ε, και για να το επιτύχουμε αυτό θα εξυπηρετούσε πολύ η συμπερίληψη αυτού του μικρού νησιωτικού κράτους στην ε, Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για να προχωρήσουμε με την ε, ε, δουλειά που κάνουμε σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ, David. Ναι. Θα συνεχίσω ακριβώς στη γραμμή των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι όντως πολύ σημαντικό να κυρωθεί η συμμετοχή σε αυτή πολύ περιορισμένη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης η Σαμόα, ε, αλλά πρέπει και να τονίσουμε ότι θέλουμε μια πλήρη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης για όλες τις χώρες του ειρηνικού, με ιδιαίτερη έμφαση στο εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη, στο ε, δίκαιο εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και θα συμφωνήσω επίσης ότι πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους κεφάλαια ε, σε όλε τι οικονομικές, συμφωνίες οικονομικής εταιρική σχέση. Αλλά ταυτόχρονα και ο Πρεσβευτή Σαμό μα είπε ότι κάθε χώρα έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί ε, είναι καλό το ότι η ΣΑΜΟ είναι διατεθειμένη να ε, ενσωματωθεί και δεδομένου ότι από την 1η Ιανουαρίου χάνει τα οικονομικά της, τα εμπορικά της προνόμια, δεν πρέπει να την αφήσουμε να την εγκαταλείψουμε. Ο Ρόμπερτ Λούι Στίβενσον, σπουδαίο Σκοτσέζο συγγραφέας, όχι μόνο του Dr. Jekyll, Mr. Hyde, αλλά και του νησιού των θησαυρών, της νήσου των θησαυρών, έχει περάσει μεγάλο μέρο, είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του στη Σαμόα, εκεί έζησε και μας την περιέγραψε. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι ένα νησί το οποίο αξίζει να το στηρίξουμε με την ε, πρόσβαση στην ε, ευρωπαϊκή αγορά και όπως είπε και ο σκιώδης μας δεν είναι μέρος του προβλήματος του, της, ε, των, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα Ισαμόα, αλλά θύμα των βιομηχανικών εκπομπών άλλων κρατών και δεν πρέπει να τιμωρηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Πρέσβη για την παρουσία του εδώ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση του θέματος για σήμερα και η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ορίζεται στις 6 Νοεμβρίου. Okay. On the next meeting, we will have yes, first the draft report and then. Ναι, τώρα θα περιμένουμε πρώτα το, πρώτο, το, το σχέδιο της έκθεσης και μετά θα προσδορίσουμε τον, την ε, προθεσμία για την καταθέση των τροπολογιών. Σας ευχαριστώ πολύ και περνώ στο σημείο 16 της έκθεση ελέγχου των ε, οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των χρηματοπιστωτικών και κυρίως των εξωτερικών χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων ο κύριος Ντάρτμουθ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Δεν βλέπω τόσο πολλούς συναδέλφους. Έστω ε, πνεύματι ελπίζω να μας παρακολουθούν. Ξεκινώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μια ιστορική προοπτική. ΕΤΕΠ. Εγκαθιδρύθηκε με τη συνθήκη της Ρώμης του 1958 ε, ως τράπεζα δανεισμού μακροχρόνιου Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πρώτα απ' όλα είναι τράπεζα. Δηλαδή πρέπει να δρά υπό τις βασικές και κοινέ αρχές τις τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές ή ε, εμπορικού κέρδους. Και αν δεν το πράξει αυτό μπορεί να μας φανεί ακριβώς αλμυρός ο λογαριασμός. Και επίση θα ήθελα να σημειώσω, να σημειώσω ότι είναι πολλέ οι τράπεζε που έχουν προβλήματα, όχι όμω η ΕΤΕΠ. Και δεν θέλω να στεναχωρήσω τον πρόεδρό μα, αλλά η Deutsche Bank ε, συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών που έχουν τα πολύ σοβαρά προβλήματα. Έχει λοιπόν να κάνει με δανεισμό κεφαλαίων από τι κεφαλαιοχικέ αγορέ, με τον οποίο χρηματοδοτεί τα έργα ε, από πλευρά τη. Είναι πολύ σημαντική και μεγάλη τράπεζα με κεφάλαιο 243 δισεκατομμύρια ευρώ ε, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι μεγαλύτεροι μέτοχοι Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ενωμένο Βασίλειο έχουν 16,11% μερίδιο έκαστος με 39 δισεκατομμύρια και άνω ευρώ κεφάλαιο και πρέπει να επισημάνουμε ότι ακόμα και η Σλοβακία με 0,25% μερίδιο ε, αντιστοιχεί ισοδυναμή σε 600 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για πολλά, πολλά χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει δημοσιονομική εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να καλύψει τους κινδύνους τους. Βέβαια, ο κίνδυνος εδώ θα ήταν αυτός του ηθικής ε, ζημίας, του ηθικού κινδύνου με συγχωρείτε για τη λέξη hazard, αλλά εγώ που είμαι της ε, Chelsea υπουργο, ε, οπαδός, έχω ένα θέμα με την προφορά της λέξης Αζάχ. Ε, ας το ξαναπώ λοιπόν, moral hazard. Ε, ηθικός κίνδυνος λοιπόν. Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί να έχει απεριόριστα δυνάμει ε, κονδύλια στη διάθεσή της τράπεζα, κινδυνεύει να αναλάβει πιο ε, ε, πιο επισφαλή έργα, πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Επίσης, 25% της χρηματοδότησής της και περισσότερο ε, αφορά το περιβάλλον, να αναμένεται μέχρι το 2020 να ανέλθει στο 35%. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η χρηματοδότηση, ο δανεισμός που έχει να κάνει με έργα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής επι, επαναλαμβάνεται ή επικαλύπτεται με άλλες αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις και αυτό είναι μία από τις συστάσεις της ε, ε, γνωμοδότησής μου να επανεξεταστεί αυτό. Επίσης, ο δανεισμός της ΕΤΕΠ προς την Τουρκία ιδιαίτερος, αλλά και χώρες της ε, εταιρική σχέση με την ε, Συμφωνία Λίβανο, Ιορδανία, Αίγυπτο, με αρκετά υψηλά ποσά που θεωρούν ότι αφορούν χώρες που έχουν κριθεί από την ε, Transparency International, τη Διεθνή Διαφάνεια, ως ε, μάλλον ε, αδιαφανείς και διεφθαρμένες, θα πρέπει να επανεξεταστούν. Ένα περιθωριακό σχόλιο για τον δανεισμό σε σχέση με το περιβάλλον μπορεί να έκανα, αλλά θα ήθελα επίσης να συμπληρώσω ότι τα δάνεια της ΕΤΕΠ έχουν χρησιμοποιηθεί από ορισμένε εταιρείε μέσα στο σκάνδαλο των εκπομπών, όπως της Volkswagen παραδείγματι, που σημαίνει ότι μπορεί η ΕΤΕΠ να έχει χρηματοδοτήσει δραστηριότητες και αντιδιοντολογικές αλλά και παράνομες ακόμα. Στη γνωμοδότηση επίσης επισημαίνουμε ότι η ΕΤΕΠ θα πρέπει να ενισχύσει τη διαφάνειά της. Όχι μόνο έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και τη λογοδοσία προς τα Εθνικά Κοινοβούλια των κρατών μελών, των μελών τη, γιατί είναι απολύτω λογικό να μπορούν να ελέγχουν περισσότερο τι δραστηριότητέ της στα Εθνικά Κοινοβούλια. Κάποια ειδική ρύθμιση πρέπει να προβλεφθεί για τον μεγάλο μέτοχο Ηνωμένο Βασίλειο ε, και Μια και δεν έχω πολύ χρόνο. Θα θέλω απλώ να επισημάνω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ο όγκο τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, όπω είπα, πάνω από 600 δισεκατομμύρια και δεν μπορεί να παραγνωριστεί αυτό και στο μέλλον. Επίσης, η προσήλωση σε ε, πρακτικές των κοινών εμπορικών τραπεζών, της κοινή τραπεζικής ε, λογικής είναι πολύ σημαντική, πρέπει να συνεχιστεί. Και αυτά, κάποια άλλα σχόλια τα αφήνω για το τέλος της συζήτησης. Ευχαριστώ. Σκιώδης, ε, πρώτος ο κύριος Σάινφελτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. εξαντλητική η παρουσίαση αυτή. Κάλυψε ένα ευρύτατο φάσμα πολλών και διαφόρων θεμάτων και μπορεί να έχουμε κάποιες αφιβολίες και αυτές τις ανέφερε. Η έκθεση αυτή είναι αιτήσια αξιολόγηση αλλά επίκειται και η 60η επέτειος της ΕΤΕΠ και ίσως είναι αυτή μια ευκαιρία να δούμε την ευρύτερη εικόνα της αποτελεσματικότητας και της ε, δράσης ε, της τράπεζας αυτής. Τρεις είναι οι βασικοί στόχοι της. Να δημιουργεί οικονομική ανάπτυξη και επασχόληση, θέση εργασίας δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά δεύτερο λόγο να υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη συμπεριλαμβανομένης και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και αυτό μας ενδιαφέρει εμάς στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου που είναι υποστήριξη της ευρωπαϊκής πολιτικής και πρόθεση εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ήταν ο τρίτο στόχο. Ιδιαίτερα ο τελευταίος λοιπόν μα ενδιαφέρει εμά και θα πρέπει να τον έχουμε υπόψη μα στι εκθέσει μα. ο προϋπολογισμός χωρίζεται σε διάφορους τίτλους. Και έχει σημασία αυτό ε, αν εξετάζουμε τις ενδοενωσιακές δράσεις της τράπεζας ή τις δράσεις της εκτός. Αν δούμε το 10% του προϋπολογισμού της τράπεζας να διαιρείται δια 150 κράτη στον κόσμο, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μικρά ποσά και πώς μπορούμε να επιτύχουμε με τέτοια μικρά ποσά τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός αυτής. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει κατά την άποψή μου. Επόμενο θέμα. Αρκούν οι επενδύσεις αυτές για να επιτύχουμε τους πολύ σημαντικούς στόχους στους οποίους έχουμε θέσει. Παράδειγμα, η Ευρώπη 2020 Αυτό έχει σημασία. Και πάλι ε, όταν εξετάζουμε τη δράση της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Απαιδήσεων εκτός της Ένωσης. Έχει σημασία και στα πλαίσια του Brexit. Δεν αφορά μόνο την παρούσα έκθεση φυσικά, είναι προφανώς σχετικό λόγω της συμμετοχής οικονομικής του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά θα επηρεάσει και ολόκληρο το σύστημα ε, λόγω των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει προς την ΕΤΕΠΗ, η Μεγάλη Βρετανία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να δούμε και τις αρχές που διέπουν τη δράση της τράπεζας. Αυτή θα πρέπει να δρά περιφερειακά ή εγκάρσια, οριζόντια γενικά. Υπάρχει και ένας άλλος τομέας που θα πρέπει να μας απασχολήσει και να εξετάσουμε Και αυτό είναι, θα πρέπει να βασίζεται η τράπεζα σε εμπορικές αρχές ή θα ε, ε, πρέπει να είναι μια οργάνωση παροχής βοήθειας και αρρωγής. Είναι περίπλοκη στη δομή της ΜΕΝ, αλλά παραμένει τράπεζα. Είναι ένα εμπορικό ίδρυμα πιστοτικό, το οποίο διέπεται από ε, το αστικό δίκαιο, αλλά έχει και μια ε, λειτουργία που έχει να κάνει με το δημόσιο δίκαιο λόγω το, της συμμετοχής των κυβερνήσεων. Και ερχόμαστε τώρα στη διαφάνεια, τη διαφάνεια των αποφάσεων που λαμβάνονται έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι στόχοι προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ανέφερα έτσι λοιπόν αμέσω μέσω έξι θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν και θα κάνω σχετικά τροπολογίες για να επικεντρωθούμε σε αυτά. Η έκθεση αυτή είναι αρκετά ευσύνοπτη και δεν επεκτείνεται πάρα πολύ σε αυτά τα θέματα. Και σας ανακοινώνω ήδη από τώρα ότι θα κάνω τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Άλλη σκιώδης. Μόνο το Γιάννη Ξαντό βλέπω. Euh, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή που έκανε μια έκθεση τόσο προσωπική, τόσο κοντά στις θέσεις του. Είναι καλό να βλέπει κανείς έναν βουλευτή που δεν προσεγγίζει το θέμα τεχνοκρατικά και εκφράζει τις προσωπικές του πολιτικές θέσεις. Ήταν επίσης χαριτωμένο που έκανε το σχόλιο για την Τσέλση. και ίσως να είναι από τις ε, ομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη που έχει τους περισσότερους παίχτες από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει και σε κάτι στο Βρετανικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν, έχει Γάλλους, έχει ε, Βέλγο, έχει έναν Ισπανό. Να λοιπόν που αυτή η ε, χωνευτήρι, αυτή η συμμετοχή των Ευρωπαίων κάνει και καλό όταν πρόκειται τουλάχιστον για το ποδόσφαιρο. Ο συνάδελφος με την προφορική του παρουσίωση ξεκαθάρισε κάποια πράγματα που στην γραπτή εκθέση δεν είναι σαφή. Για παράδειγμα, όταν λέει ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε το μέρο, ποιο ποσοστό των επενδύσεων πηγαίνει για δράσεις υπέρ του κλίματος, θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι συμφωνεί με τους οικολόγους που ζητούν οι επενδύσεις της EIB, της ε, Τράπεζας Επενδύσεων, να χρησιμοποιηθούν πολύ περισσότερο για την δράση κατά το κλίμα. Θα με είχε ε, εκπλήξει κάτι τέτοιο. Εμείς θα υποβάλουμε σχετικές τροπολογίες, έτσι ώστε πράγματι μετά και από την τελευταία έκθεση για το κλίμα την προηγούμενη εβδομάδα να ενισχύσουμε τη δράση της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς, τα εκεί. Ο συνάδελφος μίλησε για moral hazard, για να ακολουθήσω και την προφορά του. Έχει δίκιο. Υπάρχει ένα θέμα και πρέπει να υπάρχουν εγγυήσει για το ενδεχόμενο αυτό. Όμως, Αναρωτιέμαι τελικά ποιος είναι ο στόχος. Είναι μήπως να απαλλαγεί κανείς από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή θέλει πραγματικά να την ενισχύσει. Γιατί. Εάν μιλούμε για χρηματοδότηση κρατών με διαφθορά, το καταλαβαίνω. Το έχουμε επισημάνει και εμείς πολλές φορές ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να προσέχει πολύ περισσότερο και να ερευνά την ποιότητα της διοίκησης των κρατών στις οποίες στέλνει βοήθεια. Αλλά εάν το ε, ε, επεκτείνει υπερβολικά κανείς αυτό το επιχείρημα, τις μισές επενδύσεις που έχει, στείλει, έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν θα έπρεπε να τις έχει κάνει. Επομένως, χρειάζεται ε, μια προσοχή. Βεβαίως πρέπει να εξετάζεται πιο, περισσότερο ενδελεχώς το ζήτημα της διαφθοράς. Εάν λοιπόν με την έκθεση αυτή ε, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μάλιστα. Εάν αντιθέτως με την έκθεση αυτή προσπαθούμε να την καταστρέψουμε, δεν θα τύχει της υποστήριξης των οικολόγων. Την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρώτα απ' όλα για το ζήτημα της εθνικής ηθικής διακινδύνευσης, moral hazard. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές, διαφορετικά εχέγγυα ανάλογα με τη δραστηριότητα για την οποία συζητούμε. Γιατί αναλαμβάνει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες η ε, Τράπεζα Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σίγουρη ότι ακολουθεί μια συντηρητική πολιτική. Θα έλεγα μάλιστα ότι σε ορισμένε περιπτώσει η Επιτροπή θα προτιμούσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να είχε αναλάβει περισσότερου κινδύνου, να είχε ε, ενισχύσει περισσότερο κάποια έργα τα οποία δεν μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα. Μπορώ λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχουν εγγυήσεις χέγγια που να επιτρέπουν ε, να περιορίζουν μάλλον το ε, πιθανότητα να αναλάβει υπερβολικούς κινδύνους. Για το ζήματα του κλίματος. Βρίσκεται και στην πρότασή μας μάλλον για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη σχετική δέσμευση και από την πλευρά της Τράπεζας Επενδύσεως. Όσον αφορά το Brexit, το είπατε και εσείς, 39,2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το συνολικό ε, μερίδιο της Ευρωπαϊκής, ε, της, του Ηνωμένου Βασιλείου. 3,5 είναι χρηματικά διαθέσιμα στην τράπεζα. Και ένα μέρος της διαπραγμάτευσης για τον Brexit με βάση το άρθρο 50 είναι πώς θα γίνει αυτή η ανάκτηση των 3,5 δισεκατομμύρια και του, ε, ε, μέχρι το 2030 και από εκεί και πέρα θα αποχωρήσει, θα, θα ανακτήσει το, το μερίδιο του το Ηνωμένο Βασίλειο πληρώνοντας τα, στη συνεισφορά του προράτα στα, διάφορες δάνεια τα οποία έχει ήδη εγκρίνει η ε, Τράπεζα Επενδύσεων. Σας ευχαριστώ. περιμένουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τελικό αποτέλεσμα της έκθεσης αυτής της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Okay. Καλώς. Ωραία. Κύριε Σιγητά μου, να κλείσουμε. Ναι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκανε μια πολύ συνεπή απόπειρα να απαντήσει σε κάποια από τα θέματα που εγώ έθιξα προηγουμένως. Δεν συμβαίνει πάντα εδώ στην Επιτροπή μας να απαντάει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα σχόλια των βουλευτών. Και πραγματικά το εκτιμώ και ήθελα να το πω. Το έχω σκεφτεί και το ε, εντυπωσιακό τώρα ε, σχετικά με την Τράπεζα Επενδύσεων ποιο είναι. Υπήρξε μια παγκόσμια μαζική τραπεζική και χρηματοπιστωτική κρίση μετά το 2009 που για να το πω ωραία και ουδέτερα πολύ μεγάλα ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατέρευσαν το EA, IG, Lehman Brothers, κινδύνευσε η Citibank και άλλες. Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που είναι κρατικό ίδρυμα κατάφερε να τα αποφύγει όλα αυτά. Και Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και τις πιστώνεται το γεγονός και ακόμα και το γεγονός ότι κινήθηκε σε πολύ συντηρητικά επίπεδα και σώθηκε. Γίνονται, ακούγονται πολλές επικρίσεις, αλλά αν χαλαρώσει την εμπορική της πρακτική, ε, αυξάνεται ο κίνδυνος να πάνε στραβά κάποια πράγματα. Ε, θα πρότεινα λοιπόν να συνεχιστεί η διαχείριση όπως δεν υπάρχει μεγάλη όρεξη εδώ να γίνει συζήτηση σε βάθος για το πώς θα πρέπει να διαρθρώνεται η τράπεζα ε, κατά περιφερειακό τρόπο όπως ισχύει σήμερα ή εγκάρσιο γενικότερα. Δεν βλέπω να τρελαίνεστε για τη συζήτηση αυτή. Οπότε ας σταματήσω εδώ και περιμένω τις γραπτές τροπολογίες σας που θα προκύψουν από αυτή μου την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. Λοιπόν, η προθεσμία για την κατάθεση των ανθρωπολογιών είναι η 15 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. 15 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα. Και ολοκληρώνεται εδώ το σημείο 16. Και πάμε στο 17 που είναι η πρώτη ψηφοφορία. 7 λεπτά διάλειμμα. Ακριβώς στις 10 είναι οι ψηφοφορίες. So, dear colleagues, ladies and gentlemen, be quiet. Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να ξανά ξεκινήσουμε. Γιατί έχουμε τώρα ψηφοφορίες ε, στο 17 περνάμε. Αλλά πριν να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή, κάνουμε μια δοκιμαστική παρακαλώ. με τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Άρχεται η ψηφοφορία. So, and the vote is closed. Λοιπόν, τέλειωσε η δοκιμαστική. okay, so can... Όλα καλά λοιπόν, εντάξει, πάμε, ψηφίζουμε, αρχίζουμε. Σημείο 17 για την κατάργηση των ασφαλιστικών δικλείδων κτλ. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37. Τροπολογία υπέρ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 Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ Against. κατά αποχές απορρίπτεται. Compromise 3 in Συμβιβαστική 3 υπέρ Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Against. Abstention. Reject. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 65 με προφορική τροπολογία. Παρακαλώ, Γιάννη Ξοντό. Ευχαριστώ. Η σημερινή διατύπωση του κειμένου ε, είναι μάλλον δυσνόητη και προτείνουμε να συμπεριληφθεί κάτι και είναι η τελευταία φορά που μπορούμε να το κάνουμε για τα κοινωνικά και τα ε, περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα πρέπει λοιπόν εκ των προτέρων να εξηγούνται και είναι τα αιτία του αθέμητου ε, ανταγωνισμού που προκύπτουν από παραβίαση της σύμβασης ΑΕΛΟ και συμφωνία του Παρισίου. Ωραία. Με αυτή την αλλαγή ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτωτο. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 κατά αποχές εγκρίνεται. Η 69 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 70 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 77 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται 78 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται 79 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται 80 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται 82 υπέρ κατά απόχες απορρίψετε.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 Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Φιέλνερ. Θέλουμε να κάνουμε την αλλαγή που βλέπετε εδώ στον κατάλογο ψηφοφορίας. Από τέτοιες διαδικασίες με τις διαδικασίες μηχανισμούς του άρθρου 14. Μάλιστα ψηφίζουμε με αυτή την τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 καταπίπτει μάλιστα η συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 13 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται και τώρα τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά σας παρακαλώ αρχίζει τώρα so one EPP is... Ένας από το ΕΛΚ υπεράριθμος, τώρα όχι. So, everybody voted. Ψηφίσατε όλοι, πέρασε. εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Συγχαρητήρια κύριε Φιέλνερ. Θέλετε να πείτε τίποτα. Ευχαριστώ. Τι κάνατε για να βγει τόσο μεγάλη ψηφοφορία, τέτοια, τέτοιο αποτέλεσμα. Μάλλον θα έχω πολύ την ψυχή μου. τώρα μπορώ να αρχίσω να διαπραγματεύομαι με το Συμβούλιο, έτσι ώστε να τελειώσει το συντομότερο το θέμα. Γιατί συμφωνούμε όλοι στο εξή. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε νέες εμπορικέ συμφωνίες. Καλό είναι να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες και να είναι σαφείς οι κανόνες που ισχύουν. Σας ζητώ λοιπόν την άδεια να αρχίσω διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Μάλιστα, ο εισηγητής μας ζητάει να του δώσουμε εντολή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 69 του κανονισμού ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ αρχή ψηφοφορία τώρα εγκρίνεται λοιπόν αρχίζουν διαπραγματεύσεις καλή τύχη η απόφαση αυτή θα ανακοινωθεί στις 22 Οκτωβρίου στην Ολομέλεια. Ωραία, θα συνεχίσουμε λοιπόν με το σημείο 18. Δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά σε ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για την 6. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σα παρακαλώ να σηκώνετε ψηλά το χέρι σας για να μην κάνουμε λάθη. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβ... Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά για τη 18. Πέρας ψηφοφορία. Να ακολουθείτε τον κατάλογο της ψηφοφορία και όχι πάντα τον κοινοβουλευτικό σας ε, αρχηγό. Ε, συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, ε, ε τμήματική ψηφορία για το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα της 28. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ξεκάθαρα. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 τμήματική. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. 31. The vote is open. And the vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική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 απορρίπτεται 16 τμήματική ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται για το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε θέλετε ψηφίστε ηλεκτρονικά για τη 17 The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά για το κείμενο που τροποποιήθηκε. Ψηφίστε παρακαλώ. And the vote is... Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Πάμε τώρα στο σημείο για την δει Σε... Μια μιλήτρια, να δούμε, γιατί δεν βλέπουμε στην οθόνη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Μπορείτε να το ανακοινώσετε, δεν το βλέπω. Ah, sorry. It doesn't function sometimes, I apologize. <laughs> no, but the touch screen is very sensitive, so it sometimes doesn't work. I apologize ζητά συγγνώμη η γραμματεία γιατί έχει μια οθόνη αφήση η οποία είναι έτσι πολύ ευαίσθητη και καμιά φορά δεν δουλεύει. Ωραία, σημείο 20 τη ημερήσης διάταξη. Ενδιάμεση έκθεση για το πολιτέ δημοσιονομικό. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, Αποχέ. Εγκρίνεται. Η 5 καταπίπτει. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Για την 9. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική... Όχι, θέλετε να ελέγξουμε για την 18. Ψηφίστε ηλεκτρονικά για την 18. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20... Ε, θέλετε να ψηφίσουν 24 ηλεκτρονικά, ψηφίστε παρακαλώ. And the vote closed. Πέρας ψηφοφορίας, απορρίφθηκε 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές δεν είμαι σίγουρος ψηφίστε ηλεκτρονικά για την 29 παρακαλώ The vote closed. απορρίπτεται 30 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. 21. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Και ξεκινώ. 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές και νομίζω ότι έχει απορριφθεί αλλά στο επαληθεύσουμε. 25 λοιπόν αρχίζει η ψηφοφορία.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 κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, επαληθεύουμε. 16. You're might right, Christoph. Okay, the vote is closed. δίκιο, Κρίστοφ, και απερίφθη. 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η προφορική 2 που όμως ε, είναι συναφής με την προφορική 1, δεν την ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Καλά, επαληθεύουμε. Για να δούμε. Ε, είδατε ότι ήταν ίσα ίσα. Αλλά περίφθη. Αλλά ήταν και πολύ ίσα ίσα. Ολόκληρη η έκθεση λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ άρχεται. Και πέρας. Εγκρίνεται με ευρύτατη πλειοψηφία και συγχαρητήρια στην Κάρολιν Γκράσβαντλ Ντερ Χάιντς. Σας ευχαριστώ πολύ. So, this is, uh, the end Και έτσι ολοκληρώνονται οι ψηφοφορίες μας. θα ακολουθήσει το σημείο 22. Θα θυμάστε ότι έχουμε αναβάλει το 23, 24, 25 και έτσι θα παρακαλέσω τον εισηγητή του 26 να είναι εδώ το ταχύτερο. be quiet. We switch now to... Συνεχίζω παρακαλώ, σημείο 22. Ομάδες παρακολούθησης ε, ΑΖΕΑΝ πρώτα. Κύριε Ντέβιτ Μάρτιν, έχετε το λόγο. Thank you, Chair. Um, it seems a long time ago. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται σαν να έχει πέρασει πολύ χρόνο, αλλά 28 Αυγούστου είχα την τιμή να προεδρεύσω τη ε, ε σχετική ομάδα ΑΖΕΑΝ που είχε ασχοληθεί με την ε, Ινδονησία 9 με 13 Ιουλίου. Είχε προηγηθεί μια συνάντηση στις Βρυξέλλες και, πριν την, ε, και τα θέματα που, τους απασχόλη, που μας απασχόλησαν ήταν δεσμολογικά κυρίως συναλλαγές σε υπηρεσίες δημόσιες προμήθειες όπου δεν έχει αναλάβει ούτε μία δέσμευση για πρόοδο η Ινδονησία και έτσι δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει ανταλλαγή προσφορών. Πρόοδο δεν έχουμε στο σύστημα επενδύσεων ούτε στο TSD, τις συζητήσεις TSD. Θέματα λεπτά όπως πρόσβαση σε φαρμακευτικά προϊόντα και SPS δεν συζητήθηκαν στο τελευταίο γύρο. Τελευταία είδηση, αλλά καλή είδηση. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπόρεσαν να βρουν λύσει σε σχέση με τη συμφωνία για το φινικέλαιο. Συμφωνία και φαίνεται ότι ήταν πολύ καλύτερο το πνεύμα, το κλίμα των συνομιλιών την τελευταία φορά. Αναμένεται την επόμενη εβδομάδα ο προσεχής γύρος, αν δεν απατώ, 15 και 16 Οκτωβρίου στην Ινδονησία. Και θα ενημερωθούμε βεβαίως πλήρως μετά. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε το Μαγκρέπ τώρα. 30 Οκτωβρίου. Αυγούστου. ξέρετε ότι είχαμε αναβάλει το θέμα του Μαρόκου για την επόμενη συνεδρία σας είχα ενημερώσει και πάω στον Καναδά τώρα. 4 Σεπτεμβρίου. Ο αναπληρωτής Δημοτάρχης ε, για τις σχέσεις ε, Κάναδα Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστοιχα των υπηρεσιών ε, που θα μας παρουσιάσουν τις συνομιλίες όπως αναπτύχθηκαν. Μάλλον μας παρουσίασαν στις 26 Οκτωβρίου, της Σεπτεμβρίου, στις 18 Οκτωβρίου έγινε η συνεδρίαση της ομάδας παρακολούθησης Είχαμε μια ενδιάμεση ομάδα για τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε με τον Ιγνάσιο Καρσία Μπεσέρ. Μπεσέρο. Για την ε, εξέλιξη της εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ηνωμένων Πολιτειών, ιδιαίτερα μετά τη συνάντηση μεταξύ των Προέδρων Γιουνκέρ και Τραμπ. Κοινή Καναδά Μεξικού αναμένεται την επόμενη εβδομάδα όπου και θα συζητήσουμε όχι δεν το λένε ακόμα πια ΕΖΕΣ το λένε ε, ναύτα το λένε ειδική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού Καναδά και οι συνέπειε αυτή τη συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης άλλη intergroup για το Μαγρέπ μάλλον ομάδα της ΣΥΝΤΑ για το Μαγρέπ ιδιαίτερα την Ινδονησία έχει οργανώσει μια επισκέψη στην Τινησία για την οποία θα ενημερωθούμε αργότερα. 26 Σεπτεμβρίου είχαμε την ομάδα παρακολούθηση για την Αυστραλία. Ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο της Αυστραλιανής Γερουσίας. Αυτά για τις ομάδες παρακολουθήσεων. Now the rapporteur for the point ο εισηγητής για το σημείο 26 όμως δεν είναι εδώ. Έχει κανείς καμιά ιδέα, θα έρθει ο εισηγητής μας για την ε, Κεντρική Αμερική. Ε? Okay, good. So perhaps somebody can call uh, Για να του τηλεφωνήσει κανείς, του Ράιμαρ. <laughs> να σπεύσει. 2.27. Και περνούμε στο σημείο 27. Α, α, α, εντάξει. Δεν είχα να καταλάβει ότι εσείς αναλαμβάνετε. Επομένως... Ο Άντι, εισηγητής κύριος Χάνσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο εισηγητή μου μου έδωσε να σας διαβάσω τώρα ένα σημείωμα. Αυτά που θα έλεγε ο ίδιο. Το 2005 κυρώθηκε η Συμφωνία Σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική και το Κοινοβούλιο συμφώνησε. Από τον Αύγουστο του 2013 προσωρινά εφαρμόζεται το εμπορικό σκέλος. Ήταν η πρώτη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ δύο ε, υπήρων πολιτικό διάλογο και συνεργασία έχουμε ως κύρια στοιχεία, ιδιαίτερα στην πολιτική, την αναπτυξιακή και το τρίτο είναι το εμπόριο. Η Συμφωνία Σύνδεσης θα διευκολύνει την περιφερειακή ολοκλήρωση και θα ενισχύσει στην Κεντρική Αμερική ε, τις εξελίξεις. Παρά τις αρνητικές τάσεις ε, στην ε, Αμερική, είναι δυναμικό το εμπόριο που έχουμε και οι ροές. Στην Κεντρική Αμερική ήταν πολύ αρνητικό το γεγονός ότι είχε φύγει ένας μεγάλος ε, προμηθευτής εξαρτημάτων ηλεκτρονικών. Ε, Και επίσης έχουμε εξαγωγές καφέ από εκεί. Αλλά μέχρι σήμερα ούτε η Κεντρική Αμερική ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν είναι σε θέση να εξαντλήσουν τις ποσοστώσεις των εμπορευμάτων που προβλέπεται και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα αρχίζει ο εξυγχρονισμός και η διαφοροποίηση των εξαγωγών από την Κεντρική Αμερική. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις για την υγεία και φυτοϊγειονομικές που βλέπουμε να έχουν γίνει πρόοδοι, ε, ιδιαίτερα για το γάλα για τα προϊόντα, τα γαλακτοκομικά. Για την ανάπτυξη ε, όμως τη βιώσιμη και τη σχέση με το εμπόριο δεν έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή τα συμβαλώμενα μέρη ε, κάνουν ε, διαδικασίες και ενέργειες για να εγκριθεί το πρωτόκολλο που συμπεριλαμβάνει και την Κροατία στη Συμφωνία ε, Σύνδεσης. Η έκθεση λοιπόν για θέλει να εφαρμόζεται απρόσκοπτα η συμφωνία αυτή και οι εκτελεστικές διατάξεις να επικυροποιηθούν και να ενημερωθούν ε, και να συνεχιστούν οι προσπάθειες να εφαρμόζεται σωστά η ε, συμφωνία. Υπάρχουν εκεί και στοιχεία χρήσιμα για τις επενδύσεις και αριθμητικά στοιχεία. Εκτός αυτού θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το πρόγραμμα, το πρόβλημα μάλλον, ε, της επιβολής ειδικών φορών κατανάλωσης στα υνοπνευματόδια από πλευράς Κώστα-Ρίκα και η προστασία των γεωγραφικών ε, ε, ενδείξεων γεωγραφικής προέλευσης. Θα πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενισχύονται για να εντείνουν τις συναλλαγές μεταξύ τους, να συμμετέχουν και να έχουν όφελος από τη Συμφωνία Σύνδεσης. Κοινωνικός διάλογος και η υποπτία της εργασίας επίσης πρέπει να ενισχυθούν. Τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής που ε, έχουν εισαγάγει διακρίσεις κατά των συνδικάτων και των αυτοχθόνων λαών θα πρέπει να τερματίσουν αυτή τη συντακτική και να προχωρήσουν στην απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση για να εφαρμόζονται σωστά οι συμφωνίες αυτές. Θα πρέπει να υπάρχει η ε, ελευθερία του συνεταιρίζεστε, του συνδικαλίζεστε, ε, συλλογικές διαπραγματεύσεις για τις αμοιβέ των εργαζομένων και απαγόρευση της παιδικής εργασίας. Όλα αυτά ε, είναι πάρα πολύ κομβικά και σημαντικά σε κάποιες χώρες Κεντρικής Αμερικής και υπάρχει κίνδυνος αποσταθεροποίησης ολόκληρης της περιοχής. Αυστρία, Βέλγιο, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να ε, κληθούν επιμόνως να κυρώσουν τη Συμφωνία Σύνδεσης. Χαιρόμαστε ο εισηγητή για τη συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές. Από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι 16 ε, Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα και η ψηφοφορία στην Ίντα θα γίνει στις 3 Νοεμβρίου και στην ε, Ολομέλεια, ή Δεκεμβρίου και στην Ολομέλεια θα πάει στις 14 του Γενάρη. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα σκιώδεις συγγητές. Ο Ντέιβιτ Μάρτιν που δεν είναι η συγγήτρια των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άλλαξε το πρόγραμμα και γι' αυτό ίσως κάποιοι συνάδελφοι να μην έχουν προλάβει άλλα θέματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική του ε, έκθεση, αντικαθιστώ την που δεν πρόλαβε λοιπόν εξαιτία αυτή τη αλλαγή μας δίνει τη δυνατότητα αυτή η συζήτηση να ενισχύσουμε την εμπορική μας ε, συνεργασία με την ε, Κεντρική Αμερική επί τη βάση κανόνων. Συμφωνεί ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν προβλέψεις θα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί μάλλον προβλέψει για μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το ζήτημα του φύλου και για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Είναι κακό το ότι δεν έγινε αυτό και θα πρέπει επίσης να οριστούν σημεία επαφή. Προ την Επιτροπή. Θα θέλαμε να είναι πιο λεπτομεριακή η αξιολόγηση της συμφωνίας. Δεν έγινε πλήρης χρήση των προτιμησιακών καθεστώτων και των δασμών από την πλευρά των Ευρωπαίων εμπορευομένων σε σχέση με τους κεντροαμερικανούς ομολόγους τους. Υποστηρίζει τον μηχανισμό για τον σταθεροποίηση των τιμών της μπανάνας και τις προβλέψεις για τα υνοπνευματόδη. Θα, προσπαθεί, θα υποβάλει όμως ορισμένες τροπολογίες για να γίνει η έκθεση πιο φιλόδοξη και πιο ξεκάθαρη. Πρώτα απ' όλα, θα τονίσει τη συμμαχία που έχει η ενίσχυση της συνεργασίας με την Κεντρική Αμερική, έτσι ώστε να προστατευτεί το πολυμερές σύστημα διεθνούς εμπορίου, εν ώψη και της μεταρρύθμισης του ΠΟΕ, να έχουμε περισσότερες συγκεκριμένες προβλέψεις για την βιώσιμη ανάπτυξη ΔΗ και να αναφέρουμε ρητά το ρόλο που πρέπει να παίζει η κοινωνία των πολιτών. Οι αντίστοιχες ομάδες θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες, να έχουν τους πόρους που χρειάζονται και να μπορούν να καλύψουν το σύνολο της ε, συμφωνίας. Επίσης, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας τη διάσταση του φύλου και να έχουμε στατιστικά στοιχεία φύλο για να κάνουμε αξιολόγηση. Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο σεβασμός της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι προϋπόθεση για να συνεχίζεται αυτή η εμπορική συμφωνία, να εφαρμόζεται και κλείνει λέγοντα σήμα ότι προσβλέπει σε μια επικοδομητική συνεργασία με του υπόλοιπου σκιώδει και τον εισηγητή. Κύριο Λάγκη, ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο συνάδελφο το λόγο. Με την ευκαιρία λοιπόν θα ήθελα να καλωσορίσω τους εκπροσώπους από τις πρεσβείες χωρών της Κεντρικής Αμερικής που παρευρίσκονται στη συνεδρίασή μας. Καλώς ήρθατε. Θα δώσω το λόγο στον γνώριμο μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό, τον κύριο Γιώργενσον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας για το θέμα αυτό. Όπως και με την Συμφωνία για την Κολομβία και το Περού, η οποία ξεκίνησε να εφαρμόζεται περίπου την ίδια εποχή, πιστεύουμε ότι είναι επίκαιρη ε, η πρωτοβουλία που αναλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχουμε φτάσει σε πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας. Συνεχίζουν να εφαρμόζονται ορισμένοι δασμοί, ε, δεν έχει γίνει δηλαδή απελευθέρωση σε κάποιους τομείς, σε κάποια προϊόντα. Ε, ιδίως από την πλευρά της Κεντρικής Αμερικής κάτι τέτοιο πρόκειται να γίνεται τα επόμενα χρόνια. Επίσης δεν έχουν εκπληρωθεί πλήρως όλες οι προβλέψεις για τη λιανική πώληση, ιδίως από την πλευρά των κρατών της Κεντρικής Αμερικής. Γενικά όμως μιλώντας θα έλεγα ότι είναι μια προσαρμοσμένη συμφωνία για τις έξι χώρες της Κεντρικής Αμερικής, η κάθε μια έχει διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης και θα έλεγα ότι σε γενικέ γραμμέ έχουμε ένα καλό επίπεδο εφαρμογή και ουσιαστικέ δεσμεύσει από αυτά τα κράτη. Και σε αυτή την περίπτωση είχαμε στενή συνεργασία με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, μια συνάντηση κάθε χρόνο σχεδόν. Πέρυσι δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε. Εν μέρη για λόγους προβλημάτων ε, με το χρονοδιάγραμμα και από τις δύο μεριές. Αλλά επίσης και γιατί χρειάστηκε κάποιος χρόνος έτσι ώστε να εξετάσουμε πώς θα έπρεπε να προσαρμοστεί η συμφωνία μετά την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε όμως μια συνάντηση τον Ιούνιο που ήταν πολύ υποκοδομητική και καταλήξαμε σε πολιτική συμφωνία για το πώς θα λύσουμε αυτά τα θέματα, πώς θα προχωρήσουμε. Γύρονται τώρα τα τυπικά, οι διάφορες διατυπώσεις και με τη συνεργασία της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Σύντομα θα αποστείλουμε στο Κοινοβούλιο το προσχέδιο των αποφάσεων που χρειάζονται για να προβλεφθεί στην Συμφωνία η προσχώρηση της Κροατίας. Υπάρχουν πράγματι και ορισμένα προβλήματα με το εμπόριο, τα αναφέρετε στην έκθεσή σας. Οι ε, γεωγραφικές ενδείξεις, το προ, ε, προς, ενδείξεις προέλευσης, ιδίως με την Ικαράγουα, και τα ζητήματα διπλής ε, και τα TRQ ε, σε κάποιες περιπτώσεις προϊόντων εκτός από τα γαλακτοκομικά. Το είδαμε με τη ζάχαρη να δημιουργεί πρόβλημα. Δεν... Ε, α, Τα ρευκότας, οι μέγιστες ποσοστώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί στο βαθμό που θα περιμέναμε και ελπίζουμε να βελτιωθεί αυτό. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το εμπόριο για την ανάπτυξη. Γνωρίζουμε ότι οι χώρε αυτέ έχουν να αντιμετωπίσουν προκλήσει όσον αφορά την κυβέρνηση. Παρακολουθούμε στενά τι εξελίξει στην Ικαράγουα. Σε αυτόν τον τομέα πρέπει να γίνουν περισσότερα. Συνολικά, συμπερασματικά θα έλεγα ότι υπάρχει καλό επίπεδο εφαρμογή τη συμφωνία. υπάρχει καλή συνεργασία και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα γίνει του χρόνου και μια αξιολόγηση αντικτύπου ενδιάμεση και ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης θα δούμε προς τα που θα εξελιχθεί αυτή η συμφωνία. Το αναφέρατε κι εσείς. Ε, είναι ζητήματα αυτά τα οποία θα πρέπει να δούμε στο μέλλον πώς θα τα λύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και τον κύριο Φερνάντο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε και συμφωνώ σε μεγάλες γραμμές με αυτό που είπαν τα μέλη του ε, Κοινοβουλίου και με τον συνάδελφό μου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζετε ότι οι σχέσεις μας, οι πολιτικές με την Κεντρική Αμερική είναι, έχει, μια ιδιαιτερότητα γιατί έχουμε όσον αφορά τα, την πολιτική μια συμφωνία συνεργασίας και όσον αφορά το εμπόριο αυτή τη συμφωνία εμπορικής συνεργασίας. Ε, Εμεί ευελπιστούμε ότι θα γίνει μια επικαιροποίηση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και απευθύνουμε μια έκκληση ε, την, επαναλαμβάνω και σήμερα ότι θα χρειαστούν οι επικυρώσει από όσα κράτη-μέλη του κοινοβόλου τους δεν το έχει πράξει ακόμα έτσι ώστε να αρχίσει να εφαρμόζεται όχι μόνο στο εμπορικό τη σκέλος αυτή η συμφωνία αλλά και στο πολιτικό τη σκέλος να την αξιοποιήσουμε πλέον στο επακρό γιατί είναι πραγματικά μια συμφωνία εταιρικής σχέση. η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ασχολείται με το σκέλος το πολιτικό, κατά κύριο λόγο, όπως γνωρίζετε. Με βάση λοιπόν αυτήν την Συμφωνία Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τα κράτη αυτά και έχουμε επίσης και καλή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου στο εσωτερικό μας για να συζητούμε και να επιλύουμε όλα τα προβλήματα, όλα τα σημαντικά θέματα που ανακύπτουν στην Κεντρική Αμερική και στα κράτη αυτά. Προγραμματίζουμε όσο το δυνατόν συντομότερο να γίνει, προσπαθούμε να προγραμματίσουμε μια διάσκεψη στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και με μεγάλη προσμονή περιμένουμε την κοινοποίηση ότι έγινε επικύρωση και από αυτά τα τέσσερα κράτη-μέλη που δεν το έχουν κάνει ακόμα. Αυτά από την πλευρά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Χάνσεν. Yes, in, uh, in the... Ναι, εξ ονόματος του εισηγητού θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή και τον David Μάρτιν και τους ε, εκπροσώπους εδώ της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θα είναι σε επαφή μαζί σας ο κύριος Μπέγκε για τα περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ και όπως είπε και ο εισηγητής, προθεσμία 16 Οκτωβρίου, το απόγευμα στις 6. Και τώρα πάμε στην ad hoc αντιπροσωπεία προς την, στην Τινησία. Ε, ο ίδιος εγώ ήμουν επικεφαλής της αντιπροσωπείας που μετέβη στην Τινησία. Με την κυρία Λαλόν, τον κύριο Σίκο, κυρία Μπεκίνο, κύριο Φίσας, Λαντσίνη. Ήταν μαζί μας. να, έπρεπε λοιπόν να αξιολογηθεί η πρόοδο σε σχέση με τη συμφωνία με την Τινησία και να συζητηθούν ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από την Τινησιακή πλευρά. Ε, λίγος ο χρόνος, μια μισή μέρα. Είχαμε όμως την ευκαιρία να συναντηθούμε με πολλούς σημαντικούς εταίρους από την κυβέρνηση, από την κοινωνία των πολιτών, από διάφορους φορείς, από μη κυβερνητικές οργανώσεις και είχαμε, πιστεύω, ότι την ευκαιρία να πάρουμε το σφιγμό της χώρας, η οποία είναι σε μια φάση μετάλλαξης. Ε, ίσως δεν έχει τόση μεγάλη ε, προτεραιότητα αυτή τη στιγμή το θέμα των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, γενική πολιτική ζωή της ε, Τινησίας. Βεβαίως εμείς θέλουμε μια συμφωνία έντιμη, μια συμφωνία αμοιβαία συμφέρουσα πάντα Υποστηρίζαμε την Τινησία σε σχέση με τη συμφωνία του πλέον ευνοουμένου κράτους, ποσοστώσεις με τις ελιέ, παραδείγματι μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν το 2015 και ταυτόχρονα προσπαθούμε να καταλάβουμε και να, να υποστηρίξουμε μάλλον και σε ανάγκες εξυγχρονισμού, εκβιομηχάνηση κτλ. Αυτή τη στιγμή όμως δεν φαίνεται ο Χαράρη να, να πιέζει προς την κατεύθυνση αυτή. Η πολιτική επικαιρότητα με εκλογές ε, το 2019 δεν διευκολύνει αυτή την ε, πρόοδο και δεν αναμένουμε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Ένας από τους συναδέλφους τους εδώ παρόντες ήταν και στην αντιπροσωπεία. Όχι, κανείς. Σχόλια δεν υπάρχουν. Καλώς. Κλείνουμε και αυτό το θέμα. 28 διάφορα. Το αγαπημένο μου. Τίποτα. Α, όχι, έχετε εσείς. Όχι, Πρόεδρε, δεν ε, ήθελα να δυσκολέψω τα πράγματα και δεν νομίζω ότι είναι και δύσκολη η ερώτησή μου, μια με ερωτική μόνο ερώτηση. Απλώς η απόφασή σας για πρόορη συζήτηση στην ε, συνεδρία συγκεκρισμένων των θυρών της ε, Καμπότζης ε, με προβλημάτισε γιατί να συνέβη κάτι τέτοιο. Δηλαδή όλοι αυτοί που περίμεναν και αδειμονούσαν στα 28 κράτη-μέλη να ακούσουν τις συνεδριάσεις, το χασάν, δεν ακούσαν τα σχόλιά σας, τα δικά σας και των λοιπόν συναδέλφων. Δηλαδή και ξέρω ότι δεν ήταν και τίποτα το φοβερά απόρριτο αυτό που συζητήθηκε. Γιατί λοιπόν, ο Πρόεδρος. Καταρχήν, συμφωνώ πολύ μαζί σας. Αλλά, να ξέρετε, ήταν η πρώτη φορά που μετά αυτή την κάπως αξιοπερίεργη ή μη τι άλλο ανακοίνωση πλευράς της Επιτροπής ότι βγαίνει από τη συμφωνία τα πάντα πλήν όπλων η Καμπότζη, χωρίς καμιά παρετέρω εξήγηση, μια, ανα, μια ανακοίνωση μόνο μας έκανε η Επιτροπή και στο blog της και ε, θέλαμε αυτό να συζητηθεί ε, κάτι δίαν πριν συζητηθεί δημοσία. Χωρίς μικρόφωνο ο πρόεδρος, αλλά μάλλον κυρίως το πέρα στη συνεδρία